βιωσιμότητα. Είναι πραγματικά ενθαρρυντικό το ότι βλέπουμε το, το επίπεδο προσήλωσης των Βιετναμέζικων αρχών στην υλοποίηση της ε, συμφωνίας αυτής. Η πίεση που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ τελικά απέφερε κέρδη και αποτελέσματα. Ε, το Βιετνάμ αναθεώρησε τον ε, εργατικό του κώδικα τον Νοέμβριο. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το ελεύθερο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθε. Ε, για πρώτη φορά επιτρέπονται ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις με την κύρωση 6 από τις 8 βασικές συμβάσεις του ILO και έχει ε, ξεκάθαρο σχέδιο να κυρώσει ε, και τις υπόλοιπες δύο έως το 2021 και 2023. Αυτό ε, ε, επίσης αποδεικνύεται και από πρόσφατες έρευνες που έχει κάνει ο ίδιος ο ΑΕΛΟ όσον αφορά τι συνθήκε εργασία στο Βιετνάμ. Μπορούμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε το Βιετνάμ για να εφαρμόζει ε, αυτές τις, ε, αυτή τη νέα συμφωνία. Και όσον αφορά τις ε, δομές, τις πολιτιακές, όπως η, αναγνώριση της κοινωνίας των πολιτών ή η δημιουργία ομάδων συμβουλευτικών ομάδων. Είμαι βέβαιος ότι μέσα από του διάβλου, όπω είναι ο ετήσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα, θα μας δώσει την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε και τα εναπομείνοντα προβλήματα. Αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για έναν επικοδομητικό μελλοντικό διάλογο με το Βιετνάμ σε όλου τους τομεί. Από την άλλη πλευρά, μια αποτυχία μα να επικυρώσουμε αυτή τη συμφωνία θα μα άφηνε με πολύ λίγε ευκαιρίε και δυνατότητε για να προωθήσουμε τι μεταρρυθμίσει στο Βιετνάμ και θα υπέσκαπτε την αξιοπιστία ως εταίρου. Ευχαριστώ πολύ για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Το λόγο έχει η συνάδελφος... Βίσλερ Λίμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ψηφίσω τις δύο αυτές συμφωνίες με το Βιετνάμ γιατί είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι αποτελούν ευκαιρία και για το λαό του Βιετνάμ αλλά και για τους Ευρωπαίους. Από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Φυσικά έχουμε τεράστιες επιφυλάξεις, αλλά και εκεί πιστεύω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία ευρωπαϊκών επενδύσεων και καταστάσεων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων εκεί που υπόκεινται σε ευρωπαϊκούς κανόνες και ε, κριτήρια. Το χειρότερο είναι να αφήσουμε ανεξέλεγκτη την κατάσταση στο Βιετνάμ, γιατί με τις συμφωνίες αυτές δεσμεύεται η κυβέρνηση να δεχτεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και κυρίως την παρακολούθηση των κανόνων από κοινή επιτροπή ε, των δύο κοινοβουλίων μας. Επίσης, προβλέπει η συμφωνία, και αυτή είναι μεγάλη νίκη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει ένα μηχανισμό καταγγελιών ανεξάρτητο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και τέλος, το Βιετνάμ πρότεινε η ε, Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετέχει στο διάλογο Βιετνάμ Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό πραγματικά είναι πρωτοφανέ. και επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε μια τράπεζα διαπραγματεύσεων από την οποία συνήθω απουσιάζει. Α τα αξιοποιήσουμε όλα αυτά για να προωθήσουμε εκεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τομπέ από την Επιτροπή Ανάπτυξη. Κυρία Πρόεδρε, ε, το ελεύθερο εμπόριο είναι από τα καλύτερα εργαλεία που έχουμε για να βγάλουμε τον κόσμο από τη φτώχεια. Το έχει αποδείξει αυτό περίτρανα η ιστορία. Αλλά με τη συμφωνία αυτή δείχνουμε ότι το Βιετνάμ μπορεί να προχωρήσει στο δρόμο της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμού. Και με τη συμφωνία αυτή ελευθέρου εμπορίου βάζουμε πολύ ψηλά τις προδιαγραφές. Είναι συνολική συμφωνία και τέτοιου τύπου συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες και η Επιτροπή Ανάπτυξη χαίρεται πάρα πολύ που υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα ε, πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικά. Και επίση για το χρονοδιάγραμμα. Ε, θα πρέπει να κυρώσει ακόμα τι συμβάσει στο ΕΛΟ που εκκρεμούν και καλό τι δύο πλευρέ να αξιοποιήσουν πλήρω τι διατάξει τη συμφωνία έτσι ώστε να ενισχυθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ε, προχωρήσουν προ του στόχου βιώσιμης ανάπτυξη. Καλό επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται στενά με την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε η ανάπτυξη να αφορά και τα εργασιακά και την προστασία του περιβάλλοντο. Τέλο, η Επιτροπή Ανάπτυξη συνιστά να δώσουμε σύμφωνη γνώμη τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ από την Επιτροπή Αλίας, ο συνάδελφος Μπαρτόλο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με το Βιετνάμ προβλέπει και ένα κεφάλαιο όσον αφορά την εμπορία αλληλευτικών προϊόντων μαζί με τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ελίας ε, επεξεργαστήκαμε μια γνωμοδότηση που δεν είναι απλώς μια παθητική έγκριση τη συμφωνίας αυτής, αλλά μπορεί πραγματικά να συμβάλλει στην κοινοβουλευτική συζήτηση που γίνεται εδώ πέρα για να δώσουμε προτεραιότητα στον τομέα αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει να καταβάλει προσπάθειες στο Βιετνάμ για να ευθυγραμμιστεί με τα δικά μας τα πρότυπα. Αυτό το έκανε σε ένα βαθμό, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο μέλλον θα καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. Μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν και πολλά κενά ιδίω όσον αφορά την καταπολέμηση παράνομη αλλία. Γι' αυτό το λόγο στην Επιτροπή Αλλία ζητήσαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ πολύ αυστηρά τι προσπάθειε που πρέπει να καταβάλει το Βιετνάμ για να καταπολεμήσει την παράνομη αυτή αλία και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμα και την κόκκινη κάρτα, σε περίπτωση που το Βιετνάμ δεν συνάδει με τα πρότυπα βιώσιμη τα οποία προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους ε, του ΕΛΚ το λόγο έχει ο συνάδελφος Βίγκλερ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, αγαπητέ επίτροπε, οι διαπραγματεύσει με το Βιετνάμ ξεκίνησαν το 2012. Ολοκληρώθηκαν σε μια πρώτη φάση το 2015, στη συνέχεια ξανά άνοιξαν και οριστικοποιήθηκαν τελικά τον Ιούνιο του 2019. Σε αυτά τα 8 χρόνια ε, σημειώθηκε δραματική πρόοδος στην κοινωνία, την οικονομία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ε, βιωσιμότητα στο Βιετνάμ. Και ε, ένας, μία από τις βασικότερες δυνάμεις που οδήγησαν αυτή την αλλαγή βεβαίως ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άσκησε πίεση ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπορική και επενδυτική συμφωνία βεβαίως δίνει εμπιστοσύνη, δείχνει εμπιστοσύνη στις βιετναμεζικές ε, αρχές. Πρόσφατα μόλις ε, μάθαμε για την αλλαγή στον εργατικό κώδικα και για την δημιουργία μιας κοινή κοινοβουλευτική επιτροπής παρακολούθησης της συμφωνίας, της εφαρμογής συμφωνίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο του Βιετνάμ. Σήμερα καλούμαστε να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ή όχι στην ε, ε, συμφωνία αυτή το να αναβληθεί θα ήταν η επιλογή του 20ου αιώνα. Να πούμε δηλαδή ότι έχετε να κάνετε τα καθήκοντά σα ακόμα και ελάτε πίσω όταν έχετε κάνει τα μαθήματά σα. Όμω, στον 21ο αιώνα νομίζω ότι η στάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι διαφορετική. Αφού έχουμε δεσμευτεί απέναντι στου εταίρου μα του Βιετνάμ πρέπει να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και εγώ καλώ του συναδέλφου όπω και το ΕΛΚ να υπερψηφίσουμε τη συμφωνία αυτή για να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε τη Βιετνάμ ένα καλύτερο και πιο ελεύθερο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Ο κύριο Λάγκε εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για 2,5 λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Βίλι Μπραντ πριν από 50, χρονών, 50 χρόνια δημιούργησε την έννοια της, ε, μετα, της αλλαγής μέσω της προσέγγισης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θεωρώ ότι και εμείς μπορούμε σήμερα να συζητούμε την αλλαγή των όρων διαβίωσης ανθρώπων στο Βιετνάμ. Αυτό ακριβώς πρέπει να επιδιώξουμε μέσω των σχέσεών μας με το Βιετνάμ να βελτιώσουμε την κατάσταση και τους όρους διαβίωσης των ανθρώπων που ζουν σε αυτή τη χώρα, ιδίως με το Βιετνάμ, λόγω των ενισχυμένων ε, εμπορικών μας σχέσεων. Είμαι βέβαιος ότι αυτή τη στιγμή πολλοί από εμάς φοράμε ρούχα ε, παπούτσια από το Βιετνάμ όλα τα ε, κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες αυτή τη στιγμή που, κινούνται, που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα κατά πάσα πιθανότητα έχουν παραχθεί στο Βιετνάμ. Οπότε πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η βιομηχανική παραγωγή θα τηρεί κανόνες τόσο όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα όσο και όσον αφορά την ε, χρήση κατάλληλων χημικών νησιών. Τις κατακτήσεις αυτές όμως, κύριε Επίτροπε, τις επέβαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε σκληρές διαπραγματεύσεις και είμαι περήφανος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το γεγονός ότι καταφέραμε μέσα από την συμφωνία αυτή να ε, συμπεριλαμβάνονται πλέον και κοινωνικά πρότυπα, θεμελιώδη δικαιώματα με ένα συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα ε, ελέγχεται από την, ίδια Διεθνή Οργάνωση Εργασίας. Το ότι επιβάλαμε οι εγχώριες ε, συμβουλευτικές ομάδες, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών να στελεχωθούν από, από ανεξάρτητες ε, κοινωνικέ οργανώσει, οργανώσει κοινωνία των πολιτών, ότι διευρύνθηκαν τα όρια δραστηριοποίηση τη κοινωνία των πολιτών, το ότι καταφέραμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για πρώτη φορά στον ετήσιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετάσχει πλέον. Αυτό είναι πρωτοφανέ. και ότι θα έχουμε μια συνεργασία μεταξύ των κοινοβουλίων όσον αφορά την εφαρμογή τη συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα όσα κατακτήσαμε. Όμω, ξαναλέω και το άλλο, ότι το έργο τώρα ξεκινάει, γιατί θα συνεχίσουμε να έχουμε διαπάλη, να έχουμε τον αγώνα μπροστά μα για να βελτιώσουμε την κατάσταση διαβίωση των ίδιων των ανθρώπων του Βιετνάμ. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο ε, Κάλ Μπρόικ του Ρινιού, έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητέ ε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η Ευρώπη υπερασπίζεται το ελεύθερο εμπόριο. Αύριο μπορούμε να γράψουμε ιστορία. Είναι οι πιο φιλόδοξες εμπορικές συμφωνίες ε, που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με αναπτυσσόμενη χώρα. Θα είναι μια ε, κατάσταση αμοιβαίας ωφέλης και για τις δύο πλευρές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ είναι ήδη σημαντική εμπορική εταίρεια. Αυτό το εμπόριο θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώ, είτε υπάρξει συμφωνία είτε όχι. Αλλά με τι συμφωνίε αυτέ το εμπόριο αυτό θα είναι πιο ισότιμο, πιο προβλέψιμο, πιο βιώσιμο και που θα λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον και τους ανθρώπους. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων το Βιετνάμ βελτίωσε τα εργασιακά δικαιώματα. Έξι από τις οχτώ συμβάσεις του ILO έχουν ήδη κυρωθεί. Η παιδική εργασία έχει μειωθεί σημαντικότατα. Γνωρίζουμε ότι έχουν ακουστεί φωνές που θέλουν την αναβολή της αυριανής ψηφοφορίας καθώς οι δημοκρατικές ε, μεταρρυθμίσεις στο Βιετνάμ δεν κρίνονται επαρκείς. Παρόλα αυτά, και εμείς θεωρούμε ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει πολύ σημαντικότερη πρόοδος όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όμως πρέπει να αναρωτηθούμε σε αυτή την αίθουσα. Θέλουμε να έχουμε καλύτερη ε, δυνατότητα να προωθήσουμε τη δημοκρατία χωρί να υπάρχει μια τέτοια συμφωνία. Δεν μπορούμε να υποκρινόμαστε τους, τους, ε, ε, ότι είμαστε μεταρρυθμιστές αν δεν αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία και αυτή τη συμφωνία ως μια πλατφόρμα για την πρόθεση της ειρήνης και της δημοκρατίας. Και τα τελευταία χρόνια και κάτω από τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν διαφανεί κάποια θετικά μηνύματα. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία και ας αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα για να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Βιετνάμ από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία Λαντσίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρωτού κάνουμε οποιαδήποτε αξιολόγηση εμπορική της συμφωνίας αυτής, σας μην ξεχνάμε ότι το Βιετνάμ είναι μια χώρα όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει το μονοπόλιο της εξουσίας και δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης οι αντιφρονούντε είναι επιθύμητοι, οι κριτικέ που γίνονται πέντε στην κυβέρνηση τιμωρούνται με κάθερξη. Δεν υπάρχουν ελεύθερε συνδικαλιστικέ οργανώσει. Το κράτο ελέγχει ακόμα και τα θρησκευτικά πιστεύω. Α μην ξεχνάμε ότι πολλέ από τι δηλώσει και τι δεσμεύσει που έχει κάνει το Βιετνάμ συμφωνία αυτή είναι κενά λόγια πολύ αόριστες δηλώσεις χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και καταληκτικές ημερομονίες. Απόλυτη αντίθεση με τις θυσίε θυσίες που έχει κάνει στο περιβάλλον, για παράδειγμα, Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βιετνάμ. Ο άνθρακας συμμετέχει κατά 40% στο ενεργειακό μείγμα, ενώ προβλέπονται ακόμα να ολοκληρωθούν σύντομα 100 εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που βασίζονται στον άνθρακα. Επίσης δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις προκειμένου να καθαριστούν τα ύδατα του ποταμού Μεκόγκ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί πολύ μεγάλη απειλή καθότι από την περιοχή αυτή προέρχεται το ρύζι του Βιετνάμ σε μια ποσότητα 80.000 τόνων σε τήσια βάση. Πρόκειται για προϊόν το οποίο εισέρχεται προφανώς στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δείξει την απαραίτητη ευαισθησία στον τομέα αυτό της παραγωγής του ρυζιού. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει επίσης να δούμε ότι είναι πραγματικά αστεία η δέσμευση του Βιετνάμ όσον αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπάρξει προστασία, μάλλον ζημίες και πολύ αρνητικέ επιπτώσεις περιπτώσει δικέ μα επιχειρήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλα αυτά όταν θα ψηφίσουμε, γιατί δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θετήσουμε τι βασικέ μα αξίε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε καλούμεθα αυτή τη στιγμή να προασπίσουμε, αντί να σκεφτόμαστε μόνο το οικονομικό κέρδο, τα οικονομικά ανταλλάγματα. Ευχαριστώ. Από για λεπτά, κύριε Αφού καταψήφισα μια έκθεση συμφωνίας εχθές, ε, το Κοινοβούλιο για πρώτη φορά προσπαθεί να κάνει ένα μεγάλο σπαγκάτ από την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάμεσα σε αυτά και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με την έκθεσή σας, κυρία Βίσλερ Λίβλα, ε, για την έκθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο που ψηφίσαμε πέρσι και το Πράσινο Σύμφωνο. Το Βιετνάμ ε, είπε ότι θα τροποποιήσει τον εργατικό κώδικα, ναι, και θα κυρώσει τη συμβάση του αποκασμού Οργανισμού εργασίας. Αλλά ε, ελευθερία του συνέρχεσθε, τα ανεξάρτητα συνδικάτα κτλ. χρειάζονται μεταρρύθμιση όχι του εργατικού αλλά του ποινικού κώδικα. Αυτό ζητήσαμε ε, με αλληλογραφία που είχαμε με τις αρμόδιες αρχές της χώρας και ε, ζητήσαμε μια έκθεση της διαδικασίας κύρωση για να συνεργαστούμε με το Βιετνάμ. Αν με το διάλογο, κύριε Λάγκε, σε όταν μία κουέντον ε, έπεσαν αυτά που στείλαμε από το Βιετνάμ. Δεν μας απάντησαν καν. Ε, δεν πρόκειται να γίνουν οι ποινικέ μεταρρυθμίσεις που ζητούμε. Εμείς ε, ως κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να το δεχτούμε στο όρομα τίνος των οικονομικών συμφερόντων. Ποιον όμως κύριε Χόγκαν και κύριε Μπούρζουα, γιατί η έκθεση οικονομικής αποτίμηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι το εμπορικό μας ισοζύγιο θα χάσει. Ξυλία, ρύζι, κλωστοϊφαντουργία. Όλοι αυτοί οι κλάδοι ζητούν όπω και εμεί αναβολή τη συμφωνία. και το χειρότερο οι Βιετναμέζικέ αρχές ε, δικαιολογούν την καταπίεση των ε, ανεξάρτητων δημοσιογράφων για να μην αναφέρω τον κύριο Φαντζιγκούν ε, στο όνομα τη ελευθεροτυπία και μας ε, ε, εμπέζουν κιόλα και τον ίδιο τον πρόεδρο του κοινοβουλίου μας που είχε ζητήσει σχετικές ρυθμίσει. και για το πράσινο σύμφωνο ερχόμαστε ε, να επιβραβεύσουμε μια χώρα που είναι άναρχη και η ξυλία και η αλληλεία και η υλοτόμηση με επενδύσεις εκεί και δεν μιλάμε και για συγκρούσει συμφερόντων ενδεχόμενες που ε, ταράζουν αυτή την υπόθεση από την αρχή. Συνεχίζουμε, λε και δεν τρέχει τίποτα. Τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και εσεί συνάδελφοι, λάβατε εκκλήσει από εκατοντάδες ΜΚΟ, πολίτες, συνδικάτα, που από ό,τι φαίνεται ε, δεν εισακούεται. υποβαθμίζονται τα τελευταία χρόνια ε, τα πράγματα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάστασή τους και ήλπιζα συνάδελφοι σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι ότι θα αλλάζατε στάση σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις που έχουμε εδώ και λίγες εβδομάδες και σήμερα είμαι υποχρεωμένη να διαπιστώσω ότι η Πράσινη Συμφωνία και τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν γίνονται σεβαστά στο Κοινοβούλιο μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ζάχραντιλ από το ECR για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε μετά από οκταετής διαπραγματεύσεις είμαστε σχεδόν στο τέρμα αυτής της πορείας. Γι' αυτό επιτρέψτε μου μερικά λόγια και μιλώ ως πρώην εισηγητής για το θέμα αυτό. Όπως γνωρίζετε, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία διατέλεσα εισηγητής και ήταν πολύ καλή η διαπραγμάτευση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τήρησε απόλυτα ε, την εντολή που έλαβε από το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ του ελευθέρου εμπορίου. Τώρα που αυξάνεται όλο και περισσότερο ο προστατευτισμός, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείε αποσύρονται από διάφορες συμφωνίες. Τώρα υπάρχει ένα κενό το οποίο μπορούμε να καλύψουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται άλλη συμφωνία με καμία χώρα της περιοχής. Το Βιετνάμ έχει περισσότερα από 90 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτή τη στιγμή προεδρεύει και στην ΑΣΕΑΝ και είναι πολύ σημαντικό και για λόγους πολιτικούς και για λόγους οικονομικούς για μας να έχουμε τέτοια συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, εμείς θα βγούμε χαμένοι και αυτός που θα κερδίσει θα είναι η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο κύριος Μογαέλ από την ΚΟΕ για 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να εμβαθύνουμε μια εταιρική σχέση με το Βιετνάμ. Βεβαίως, συμφωνούμε όλοι. Αυτό περνάει απαραίτητα από μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών. Ε, λοιπόν, όχι. Αυτή είναι η ζήτηση. Εσείς έχετε τη μαγική ιδεολογία ότι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών είναι πανάκια. Ε, δεν ισχύει. Δεν συμμερίζομαι καταρχάς την αισιοδοξία ότι είναι αμοιβαία υποφελής αυτή η συμφωνία που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 30 δις έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο με το Βιετνάμ και 40 χρόνια, ε, σε 10 χρόνια θα γίνουν 40 δις λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος θα την πληρώσει, οι Ευρωπαίοι που εργάζονται στους πιο ευάλωτους τομείς, στην κλωστοεφαντοργία. Για να γίνει το Βιετνάμ ε, το μεγάλο εργοστάσιο του κόσμου θα κάνουμε μετακαταστάσεις. Λέτε θα κερδίσουν οι Βιετναμέζοι οι εργαζόμενοι γιατί θα ε, εστερνιστούν τους κανόνες του ILO. Μα κοιτάξτε ε, τι έγινε στην Νότια Κορέα. Μας έταξαν λαγούς με πετραχίλια τα οποία δεν είδαμε ποτέ. Υποκρισία είναι αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να πούμε σήμερα ότι ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μας η κυβέρνηση του Βιετνάμ. Το αντίθετο. Ε, 176 είναι η θέση του Βιετνάμ για την ελευθερία του τύπου από 180 παγκοσμίω. Ε, απίστευτη διγλωσία. Ε, ψηφίζουμε τη νέα πράσινη συμφωνία, την έκτακτη ανάγκη για το περιβάλλον και από την άλλη τύχε Γιάννη τύχα πάντα, συμφωνία Ελευθερωση συναλλαγών, τοκτόνα που δεν προστατεύει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μα δίνει την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα προτιμάει το εμπόριο απέναντι σε θεμελιώδεις αξίες που κανονικά θα έπρεπε όλους να μας εμπνέουν σε αυτό το ε, ημικύκλιο. Ολοκληρώνεται εδώ κατάλογο των ομιλητών εξ των πολιτικών ομάδων και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι πρέπει να τηρείτε και το χρόνο σας. Η κυρία Μπεγκίν έχει το λόγο για τρία λεπτά. Παρακαλώ. Σα ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, πριν από τρία χρόνια όταν ψηφίσαμε το ψήφισμά μου για μια εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε τότε ιδιαίτερα η χειρά να έχει περισσότερες συμφωνίες με χώρε υψηλή οικονομικής ανάπτυξης. Εισακούστηκε επιθυμία αυτή. Το Βιετνάμ είναι ο νέος ασιατικός τίγρης. Με ένα ΕΠ το οποίο αυξάνεται κατά 7% το χρόνο είναι μια χώρα η οποία γίνεται όλο και πιο πλούσια και η οποία αυξάνει συνεπώς τη ζήτησή της για προϊόντα υψηλής προστιθέμενης προστιθέμενη αξία, τα δικά μα ουσιαστικά προϊόντα, αυτά τα οποία παράγουμε εδώ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τη συμφωνία θα εκμηδενιστούν οι τελειωνιακοί δεσμοί για τα προϊόντα αυτά, αλλά και για άλλα προϊόντα. Και α μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι δεσμοί όπω για το τυρί, για το κρασί, για παράδειγμα, φτάνουν σήμερα ακόμα και το 50%. Για να μιλήσω για τα αυτοκίνητα, όπου έχουμε τελειωνιακού δασμού στι τάξει του 80%. Η συμφωνία αυτή επίση αναγνωρίζει 69 ε, γεωγραφικές ενδείξεις και προστατευόμενες ονομασίες. Πάρα πολλές από αυτές είναι ιταλικές. Ιδίως για την Ιταλία οι εμπορικές αλλαγές συνεχώς αυξάνονται. Ήδη οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 12% μόνο και μόνο πέρυσι. Περισσότερες εξαγωγές και εισαγωγές που φτάνουν τα 3,7 δισεκατομμύρια μεταξύ Ιταλίας και Βιετνάμ. Το Βιετνάμ λοιπόν γίνει το πρώτος και σημαντικότερος εταίρος για την Ιταλία όσον αφορά τι χώρες Άζιαν. Και βέβαια τα ποσοστά αυτά θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο χάρη στην πολύ υψηλή ζήτηση που υπάρχει ιταλικά προϊόντα. Πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα προϊόντα υψηλής ραπτικής, 65 εκατομμύρια όσον αφορά τα τρόφιμα, περίπου μισό δισεκατομμύριο όσον αφορά τη μηχανή. Είναι σαφώ επωφελή λοιπόν η σχέση αυτή η εμπορική που έχουμε με το Βιετνάμ και θα πρέπει να ταχθούμε υπέρ των δύο αυτών εκθέσεων. Υπάρχει όμω ένα πρόβλημα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν παρουσιάζει πρόοδο. Και υπάρχουν ορισμένε σχετικέ μεταρρυθμίσει οι οποίε όμω ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί από το Βιετνάμ. Συμφωνώ λοιπόν με του συναδέλφου ότι θα φέρει μεγαλύτερη ευημερία η συμφωνία αυτή, ότι θα βελτιώσει και θα βοηθήσει να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία αυτή. Θα ζητούσα όμω από του συναδέλφου να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε τον απαραίτητο χρόνο στου φίλου από το Βιετνάμ να ολοκληρώσουν τι δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει που οι ίδιοι ξεκίνησαν και κατά αυτόν τον τρόπο το Βιετνάμ θα καταφέρει να απελευθερώσει τους αντιφρονούντες, τους αντιρρησίες συνείδησης και θα καταφέρει κατά αυτόν τον τρόπο επίσης να εφαρμόσει όλες τις συμβάσεις της ε, διεθνούς, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας όσον αφορά τους ε, εργαζόμενους. Είναι μια χώρα φίλου. είμαι σίγουρος ότι, σίγουρο ότι η συμφωνία αυτή θα εφαρμοστεί το στομότερο δυνατό, αλλά θα πρέπει να επιτρέψουμε στο Βιετνάμ περισσότερο χρόνο για να κάνει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Ο κύριος Χάντζεν, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ο κανόνα του ισχυρού τώρα διέπει τα εμπορικά τον 21ο αιώνα. Αύριο θα έχουμε την ιστορική ευκαιρία να του αποδείξουμε το αντίθετο. Α δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι η δέσμευσή μα υπέρ του δίκαιου εμπορίου βασίζεται σε αφήξει κανόνε ανεξαρτήτω του μεγέθου ε, του εταίρου. Εμεί ε, ξέρουμε ότι το Βιετνάμ είναι αναπτυσσόμενη χώρα και προφανώ έχει δρόμο μπροστά του για να εξυγχρονίσει την οικονομία, το περιβάλλον και τα κοινωνικά. Αλλά η κύρωση αυτής της συμφωνίας δεν σημαίνει ε, όπως τόνισε σωστά ο πρόεδρος Λάγκε, ότι θα τερματιστεί η συζήτηση. Δεν πρόκειται να εθελοτυφλούμε ως προς την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ και κυρίως δεν πρόκειται για λευκή επιταγή που δίνουμε στην κυβέρνηση της χώρας. Κατά τα άλλα, ο πρόεδρος ε, σας όλοι αύριο ε, θα μάλλον σήμερα θα συναντηθεί με τον αρμόδιο υφυπουργό του Βιετνάμ. 45 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, 30 χρόνια μετά την έναρξη διπλωματικών σχέσεων με τη χώρα, κυρίε και κύριοι, υποστηρίζω να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας και ε, θα εντείνουμε έτσι τη συνεργασία μας και τη συζήτηση με του Βιετναμέζου, αυτή τη φορά με πραγματικού ε, μοχλού αξιόπιστου. Ε, η κοινή επιτροπή ζήτησε και πέτυχε από το Κοινοβούλιο μάλλον που ζήτησε και πέτυχε το Κοινοβούλιο, θα μας επιτρέψει ε, να ε, προωθήσουμε τη βελτίωση της ζωής όλων των Βιετναμέζων. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τόγια, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας ε, και για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την Ιταλική οικονομία και τις Ιταλικές εξαγωγές και για την ίδια τη χώρα για να κάνει ένα άλμα για την ανάπτυξή τους. Το συνειδητοποιούμε αυτό και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγον, αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε. Η κατάσταση είναι ακόμα πάρα πολύ κρίσιμη στη χώρα αυτή. Κρίσιμη όσον αφορά τα ε, ε, ανθρώπινα δικαιώματα εν γέννη και όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, όσον αφορά τις πολιτικές ελευθερίες, τους κρατουμένους και ε, όσον αφορά και συνεχίζω που το επαναλαμβάνω και με εκπλήσει που δεν δίνει σημασία ούτε καν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, μπορώ να έχω την προσοχή σας. Μπορώ να έχω την, επιτροπή, την προσοχή σας. Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπα, θα σας γράψουμε φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά όσον αφορά και την παρέμβαση για τη συνεργασία για την ανάπτυξη. Επισημάνω το θέμα τη υποχρεωτική εργασία, τη καταναγκαστική εργασία των ε, ανηλίκων και τη συνθήκε εργασία των γυναικών, που είναι απαράδεκτο. Και όχι μόνο στο Βιετνάμ. Είναι η παγκόσμια λυσίδα αξιών που οδηγεί σε τεράστια μείωση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Σίγουρα έχουν γίνει κάποια βήματα μπροστά. Το λέω με περηφάνεια εξ ονόματο όσων διαπραγματεύτηκαν εξ ονόματο τη ομάδα μου και επέτυχαν εξαιρετικά πράγματα, αλλά πρέπει να ζητήσουμε ίσω περισσότερα για την εργασία, για τι γυναίκε, για τα παιδιά. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πάρα πολύ αυτή τη συμφωνία. Εδώ διακυβεύεται η σοβαρήτητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσων κάνουν εμπορικέ ε, διεθνεί διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε. Χάν για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το εξή. Το Βιετνάμ είναι μια κομμουνιστική χώρα, δεν είναι δημοκρατία. Και μια εμπορική συμφωνία δεν θα την κάνει η δημοκρατία μια ανοιχτή. Ωστόσο, η συμφωνία θα προωθήσει τι οικονομικέ εξελίξει, θα βγάλει τον κόσμο από τη φτώχεια, θα του δώσει περισσότερα δικαιώματα και προστασία. Ο νέο εργασιακό κώδικα προστατεύει ιδίω τι ευάλωτε ομάδε, τα συνδικάτα, θα επιτραπούν, θα υπάρχει ελευθερία του συνεταιρίζεστε, μεγαλύτερη διαφάνεια και παρακολούθηση από τη διεθνή κοινότητα σίγουρα θα είναι κάτι θετικό. Έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ ήδη με το Βιετνάμ. Δεν είναι το θέμα θέλουμε να έχουμε εμπορικέ συναλλαγέ ή όχι με τη χώρα αυτή. Θέλουμε απλά να βελτιωθούν οι συνθήκε. Γι' αυτό και πρέπει να εκπέμψουμε ένα χειρό μήνυμα συνεργασία προ όλε τι χώρε ΑΣΕΑΝ Όσε δυνάμει πιστεύουν στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηριχθούν. Αλλά όχι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να συνδυάσουν το εμπόριο με τι αξίε, όπω είναι η Κίνα, για παράδειγμα. Α στηρίξουμε λοιπόν τη συμφωνία και το λαό του Βιετνάμ, ώστε να προχωρήσει προ τα εμπρό. Ευχαριστώ. Πρώτα, ευχαριστώ. Συνάδελφε Ζουβά, έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα υποψηφίσουμε μια συμφωνία που θεωρούμε ότι δεν είναι καλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε για τη Γαλλία και δεν είναι καλή για το Βιετνάμ. Εδώ και χρόνια εμεί καταγγέλουμε την οικολογική παρα, τα οικολογικά προβλήματα εκεί. Υπογραμμίζουμε τους κινδύνους της στρατηγικής εξάρτησης όσον αφορά τις πηγές εφοδιασμού που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και που παρά από τις προσπάθειές μας δεν ελέγχουμε τίποτα πραγματικά. Και εδώ και χρόνια καταγγέλουμε επίση την παρέμβαση στα εσωτερικά μια κυρίαρχης χώρα. ο πολύ συχνά ε, δίνουμε αυτέ τι συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών. Γι' αυτό δεν υπογράφουμε αυτέ τι συνθήκε, διότι πιστεύουμε ότι ο 21ο αιώνα γυρίζει τη σελίδα των ελευθέρων συναλλαγών και τη παγκοσμιοποίησεω. Θεωρούμε ότι ο 21ο αιώνα θα είναι ο αιώνα τη μεταγκατάσταση. Θα είναι ο αιώνα τη επιδιώξεω τη βιομηχανική αυτονομία των εθνών που έχουν επίγνωση των απαιτήσεων που για την εξαρτησία του. Και πάνω απ' όλα θεωρούμε ότι ο 21ο αιώνα ε, αφορά τον οικονομικό πατριωτισμό και θέλουμε το Βιετνάμ όπω και η Ευρωπαϊκή Ένωση να εργαστούν ανεξάρτητα και για να έχουν στρατηγική ελευθερία. Σα ευχαριστώ. Η συνάδελφο Καβατσίνη έχει τώρα το λόγο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το κοινοβούλιο αποφάσισε τον Νοέμβριο ότι η Συμφωνία των Παρισίων θα πρέπει να βρίσκεται σε όλα τα κεφάλαια των εμπορικών συμφωνιών. Και αυτό το κοινοβούλιο αποφάσισε το Δεκέμβριο ότι οι εμπορικέ συμφωνίε θα πρέπει να είναι εφαρμοστέ όσον αφορά κοινωνικέ προδιαγραφέ και περιβαλλοντικέ. Και το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι στην πρώτη γραμμή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι έτοιμη να υπερψηφίσει όσον αφορά τη συμφωνία για το εμπόριο τη επενδύση στο Βιετνάμ. Στην κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινούνται στο Βιετνάμ και αριθμό των πολιτικών κατομένων όλο αυξάνεται από το 2016. Η κατάσταση είναι τέτοια που τα πολιτικά και ε, δικαιώματα παραβιάζονται ε, και η κατάσταση είναι όπου η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας δεν εμπεριέχει κανόνες κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς εφαρμόσιμους. Και όχι μόνο, και όλοι οι σοσιαδημοκράτες εδώ πίστευαν ότι αυτή και λέγαν ότι αυτή ήταν η ερυθρή γραμμή, η κόκκινη γραμμή. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου μπορεί να καταστήσει πιο βιώσιμο το εμπόριο και πιο, καλό για το, πιο καλές συμφωνίες μπορούμε να έχουμε για το κλίμα. Συνάδελφοι, γελιοποιούμεθα εάν Αφού τα λέμε αυτά, στην πρώτη ευκαιρία υποχωρούμε και αφήνουμε να περάσει μια εμπορική συμφωνία που δεν ανταποκρίνεται στι επιταγέ πράσινη συμφωνία. Σα παροτρύνω σήμερα να πείτε όχι σε αυτή τη συμφωνία. Α ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναδιαπραγματευτεί και να ευχαριστηθεί η συμφωνία του με το Βιετνάμ με την πράσινη συμφωνία και να στείλουμε ισχυρό μήνυμα προ την βιετναμική κυβέρνηση να βελτιώσει την καταστροφική κατάσταση ανθρώπινα δικαιώματα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία. Πριν και όχι μετά. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ και θα παρακαλέσω τους συναδέλφους αν θέλετε να συζητήσετε κάτι. Όχι τόσο υψηλόφωνα παρακαλώ. Αγιλάρ ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι η συνολικά εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ θα ωφελήσει πολλού ε, τομεί ε, ε, τη ευρωπαϊκή οικονομία, τυρί, βόλιο κρέα, τρόφιμα γενικά. Όμω, είναι λυπηρό το γεγονό ότι για μια ακόμη φορά η Κομισιόν δεν προστατεύει έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι το ρύζι. Ε, το Βιετνάμ έχει τι πιο χαμηλέ τιμέ από όλη την Ασιατική Ήπειρο προ το ρύζι... και ανταγωνίζεται με την Ιταλία και την Ισπανία. Η οριζοπαραγωγή στην Ισπανία είναι αγανακτισμένη με αυτό το νέο συμβιβασμό που θα επηρεάσει ένα τομέα που ήδη βρίσκεται σε κρίση. Το έλλειμμα παραγωγή ρυζιού δεν σημαίνει ότι το άνοιγμα συνόρων δεν θα προκαλέσει και ανεπανόρθωτε ζημίε στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν καταλαβαίνω γιατί. Αφού υπάρχει η ρήτρα διαφύλαξη που εφαρμόστηκε στι αρχέ του 2019 με τη Μιανμάρ και την Καμπότζη, Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει τα ίδια λάθη και δεν αξιολογεί τι επίπτωση θα έχουν οι εισαγωγές αυτές στην ευρωπαϊκή αγορά και σε ένα τόσο ευαίσθητο πράγμα όπως το ρύζι. Οι οριζοπαραγωγοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να δερματίσουν. Περιβαλλοντική ποιότητα, γεωγραφική ένδειξη ε, και θα πρέπει να γίνουν μελέτες αντικτύπου, να γίνουν ε, τα απαραίτητα. Διακόπτεται η ομιλήτρια από την Πρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύντσιτς για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή πρέπει να απορριφθεί για πολλού λόγου. Ένα από τα πράγματα που πρέπει να πούμε ότι αυτή η συμφωνία, μάλλον αυτέ οι συμφωνίε, ε, συντάχθηκαν ε, με γνώμονα τη συνεργασία. Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα. Καταρχά, η συμφωνία αυτή δίνει ε, ειδικά δικαιώματα στου επενδυτέ. Αναφέρομαι στο σύστημα επίλυση ε, διαφορών. Διότι το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο για την επίλυση αυτών των διαφορών, είναι ένα απομακρυσμένο διατητικό δικαστήριο και όχι το τοπικό δικαστήριο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε μια συμφωνία παραχώρησης, ε, όπως για παράδειγμα, που θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα στην περιοχή του Ντουμπρόβνικ, και ο ξένος επενδυτής ε, σε ένα γήπεδο γκολφ έχασε όλες τις υποθέσεις ενώπιον των ε, ε, εθνικών δικαστηρίων και προσέφυγε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο και εκεί δικαιώθηκε. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση στην οποία δίνεται δίκαιο στις επιχειρήσεις αντί για την ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Μια περιοχή λοιπόν στο Βιετνάμ που είναι πολύ φτωχή και δεν έχει πόρους ε, για να προστατέψει τα συμφέροντά της, ε, θα νιώσει το ε, αντίκτυπο όταν μια πολύ μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση θα προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της ενώπιον δυτικών δικαστηρίων που δεν ε, ενδιαφέρονται για το δίκαιο. Βάρμπορν, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε Χόγκαν, αγαπητοί συνάδελφοι, το Βιετνάμ μετά τη Σιγκαπούρη είναι ο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο ε, τη Ευρώπη στην Ανατολική Ασία και με αυτή τη συμφωνία σχεδόν όλοι οι δασμοί θα πάψουν να υφίστανται. Οπότε θα ανοίξει μία ε, εκατομμυρίων ανθρώπων νέα αγορά. Ε, αυτό σημαίνει αύξηση και της αγαροστικής δύναμης ε, και για τις 600 ε, επιχειρήσεις από το Μάλμο και από τη Βόρεια Σουηδία νέες εξαγωγικές δυνατότητες και μεγάλο δυναμικό επίσης και για όσους εισάγουν από το Βιετνάμ. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη αγορά πλέον, δεν θα είναι και τόσο εύκολο επιχειρήσεις να τα φέρουν πέρα ε, και στο Βιετνάμ που είχαμε πάει το φθινόπωρο, όποιον συναντήσαμε εκεί, ε, ανθρωπιστικέ οργανώσεις, απρασπέσεις των δικαιωμάτων, ε, οικονομικούς παράγοντε κτλ. Όλοι μα είπαν ότι θα αυξηθούν κατά 16% ε, οι εξαγωγές. Αυτό είναι πολύ καλό και για τη σουηδική ε, ανταγωνιστικότητα για τις θέσεις εργασίας. Εγώ λοιπόν θα ψηφίσω υπέρ της συμφωνίας αυτής. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος, ο συνάδελφο Γκλουξμάν για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέμε ότι έχουμε ξανά για το κλίμα. Έχουμε συμφωνήσει το πράσινο σύμφωνο εδώ και ένα μήνα μόλις και αύριο μα ζητάνε τι. Μα ζητούν να ψηφίσουμε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών παραπάνω σαν τίποτα να μην έτρεχε. Αυτή η συμφωνία, αντίθετα με τι υποσχέσει μα που είναι γραπτέ στο ψήφισμα για το Πράσινο Σύμφωνο, δεν έχει κανένα μηχανισμό περιοριστικό όσον αφορά το κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Λοιπόν, τίθεται το ερώτημα για μα και είναι απλούστατο θα δίνουμε τελικά κάποια αξία στις λέξεις που εκφράζουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Βιετνάμ ε, φυλακίζει τους ακτιβιστέ, ε, ε, τους, τους συνδικαλιστές, προασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Πάτσεντ Ντούγκ, παραδείγματο χάρη, συνελήφθη διότι μας έστειλε μια επιστολή ζητώντας να μην υπογράψουμε τη συμφωνία ως έχει αν δεν δώσετε καμία αξία στα λόγια σας, καμία ουσία, να έχετε την, τουλάχιστον, να δώσετε τουλάχιστον αξία σε αυτά που λέει εκείνο. Μην ε, τη συμφωνία του, αυτό είναι στη φυλακή γιατί μα μίλησε, αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχουν και κάποια πράγματα πέρα από το Θεό του εμπορίου. Υπάρχει το κοινό μα μέλλον, υπάρχουν οι αρχέ μα. Αύριο λοιπόν είναι ευκαιρία αυτό να το δείξουμε. Ευχαριστώ. Επόμενη Βεντρέν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος ε, οικονομικός επέτερος της χώρες ε, της ε, Δυτικοανατολικής Ασίας. Έτσι, με αυτή τη συμφωνία θα μπορέσουμε να προτατεύσουμε 175 γεωγραφικές ενδείξεις και να μπορούμε να περνάμε τα προϊόντα μας χωρίς δασμούς. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ε, και κάποιες ε, ε, νίκες που καταφέραμε να έχουμε στις επιθετικές διαπραγματεύσεις που κάναμε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πράγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε πάντα δημοσιογράφους στη φυλακή παρά τις προσπάθειές μας. Με την κύρωση λοιπόν αυτής της Διεθνούς Συμφωνίας θα πρέπει να επιμείνουμε για το σεβασμό του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εμπορική πολιτική μας πρέπει να έχει ως γνώμονα τις αξίες μας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά η κύρωση σε αυτής της συμφωνίας ε, δεν είναι αυτός σκοπός. Θα, η επιτυχία θα φανεί εάν μπορέσει να εφαρμοστεί σε ένα διεθνές πλαίσιο το οποίο είναι συνώνυμο και με εμπορικό πόλεμο. Ο Χάιντερ για ένα λεπτό. Um Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Πρόεδρε, θα ψηφίσω υπέρ αυτή τη συμφωνία. Ε, είμαι υπέρμαχο ε, του ελεύθερου εμπορίου, γιατί θεωρώ ότι φέρνει κέρδη, φέρνει ε, αμοιβαία ωφέλη και επίση είναι και ένα μοκτλό ανάπτυξη. Άρα ε, υπάρχει κάτι πολύ θετικό εδώ και στη σχέση μεταξύ Ασίας Ευρώπη. Το Βιετνάμ μια δυναμική χώρα, δυναμικό το περιβάλλον, η οικονομία από τη δεκαετία του 90 στη χώρα αυτή έχει ρυθμούς ανάπτυξης ε, σταθερά του 5%. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε ακόμη μεγάλη ε, βελτίωση, άρα και ως εξαγωγική χώρα ε, είναι πολύ ενδιαφέρον, σαν ως χώρα το Βιετνάμα. Θετικά αυτά που έχω πει μέχρι τώρα, αλλά υπάρχει και ε, αρνητική πτυχή. Οι δημοσιογράφοι που επικρίνουν οι υπερασπιστέ των δικαιωμάτων από το σαλιστικό καθεστώ κατασπιέζονται, διώκονται και πολλέ φορέ μάλιστα υπό αδιευκρίνηστε συνθήκε χάνουν τη ζωή του. Ελπίζουμε ότι με αυτή τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου και εδώ θα υπάρξει μια θετική συμβολή, να βελτιωθεί δηλαδή η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο συνάδελφο Ζαντό για 1,5 λεπτό. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, και τι δεν ακούσαμε στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ε, για τις ευρωεκλογέ παντού στην Ευρώπη. Τέρμα οι συμφωνίες ελευθέρω Εμπορία που δίνουν δικαιώματα στις πολυεθνικές εναντίον των κρατών, εναντίον της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εναντίον της ε, ε, προστασίας της δημόσιας υγείας και κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων τέρμα αυτές ε, οι συμφωνίες τις οποίες, ε, με χώρες οι οποίες συμμετέχουν στην καταστροφή του κλίματος κυρίως με την αποψήλωση και τέρμα οι συμφωνίες ε, μέσω της επίθεσης στη βιοποικιλότητα για παράδειγμα με την παράνομη αλία και επίσης τέρμα οι εμπορικοί συμφωνίες κατά της δημοκρατίας και των ατομικών ελευθεριών και ξαφνικά η πρώτη συμφωνία φτάνει και όλες οι ομάδες, οι σοσιαλδημοκράτες, οι φιλελεύθερες, το ΑΜΑΡΣ, οι συντηρητικοί όλοι υπερψηφίσετε μια συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών αντίθετη στι ε, διακηρύξει και στι δεσμεύσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Green Deal, για τι αξίε τη Ευρώπη και για την ε, ε, ρυθμισμένη παγκοσμιοποίηση. Ε, όλο τυχαίω γίνεται αυτή η συζήτηση μετά από μια συζήτηση για τον Brexit. Αλλά δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι και η ψηφοφορία για τον Brexit ήταν μια ψηφοφορία γιατί ε, εγκαταλείπουμε τις λαϊκές τάξεις εδώ για να πάμε να τις πατάξουμε σε άλλες περιοχές στην άλλη άκρη του πλανήτη χωρίς δι, ε, κοινωνικά δικαιώματα. Λίγη αξιοπρέπεια, αγαπητοί συνάδελφοι, ενώπιον των Βιετναμέζων, ενώπιον των ε, ψηφοφόρων σας απορρίψτε αυτή τη συμφωνία ελευθέρων συνολογών που δεν συνάδει σε καμία περίπτωση με τις αξίες της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιούζιτσα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δημοκρατική χώρα το Βιετνάμ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα στηρίξω τη συμφωνία για του λόγου του ότι από το 2009 το ε, Βιετνάμ ήταν 32ο ε, μεγαλύτερο ε, εισαγωγέα και πρόσφατα και ο δέκατος. Ε, υπάρχουν αλλαγές ε, που θα συμβούν με αυτή τη νέα συμφωνία. Θα βελτιωθεί και η δημοκρατία στη χώρα αυτή ή τέλο πάντων αν δεν υπάρχει θα ε, αρχίσει να αναπτύσσεται σε αυτή τη χώρα. Επίσης θα υπάρχουν οι δυνατότητες της επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που δεν βελτιώνονται οι συνθήκες. θα είναι πολύ πιο κοντά ε, το Βιετνάμ στη διεθνή κοινότητα αν βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και της δημοκρατίας στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, Ραντατσόφσκι. Εγώ θα στηρίξω τη συμφωνία αυτή. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2020 ε, συμμετείχα ε, στις Βρυξέλλες ε, σε ένα συνέδριο και εκεί γινόταν λόγος για τον Παγκλαντές και την εξαγωγή ειδών κλωστευαντουργίας και ένας εκπρόσωπος έλεγε ότι με αυτή τη συμφωνία το Μπαγκλα... θα έχανε πάρα πολλά εκατομμύρια 30 ε, δις από, την, ε, ε, από τα διαφυγόντα κέρδη. Άρα για τον Μπαγκλαντές τι σημαίνουν όλα αυτά. Χάνει ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς του. Ελπίζω οι μεγάλοι όμιλοι να μην έχουν επηρεάσει. Μιλώ για του όμιλου κλωστεβαντουρία και ειδών γιατί γνωρίζουμε πώ δουλεύουν και υπό ποιε συνθήκε παιδιά ε, σε αυτά τα εργοστάσια. Και θυμάμαι και τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Θυμάμαι το χωριό Μιλάει. Οφείλουμε κάτι πραγματικά στο Βιετνάμ, τους χρωστάμε και πρέπει να στηρίξουμε και να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία, γιατί αν δεν το κάνουμε θα ξανά πέσουν βόμβες πάνω στο λαό του Βιετνάμ. Σιμών για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, αυτή η εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ αποδεικνύει ότι μπορούμε να επιβάλλουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές μέσω εμπορικών συμφωνιών στον κόσμο. Σημαντικέ βελτιώσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων, απαγόρευση καταγκαστικής εργασία, η βελτίωση ανεξαρτήτων συνδικάτων, μηχανισμό επιβολή για τη Συμφωνία των Παρισίων που δεν θα είχαμε χωρί την συμφωνία. Τι μεγάλη επιτυχία. Συνάδελφοι από τους Πρασίνους και την Αριστερά εν γέννη είναι κατά των εμπορικών συμφωνιών και είναι κοινό στοιχείο με τους ακροδεξιούς λαϊκιστές ήρης τον παρόδο. Το ερώτημα πρέπει να απαντήσετε τώρα είναι πώς θέλετε να εφαρμόσετε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές όλο τον κόσμο μέσω των ομιλιών εδώ στο Κοινοβούλιο, μέσω διαδηλώσεων, μέσω επιστολών η μόνη ρεαλιστική προσέγγιση να προωθήσουμε την επιρροή τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο σε μια εποχή που έχει μεταβολέ γεωπολιτικέ είναι μέσω εμπορικών συμφωνιών. Εκείνοι που θα καταψηφίσουν τη συμφωνία θα πρέπει να εξηγήσουν πώ θέλουν με ρεαλιστικό τρόπο να πετύχουν του κοινού μα στόχου ενώ ταυτόχρονα θέλουν να ακολουθήσουν μια ατζέντα που απομονώνει και αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν εμπορικό εταίρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Ντάντη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, τα στοιχεία μας λένε ότι το 2018 οι εμπορικές ε, ανταλλαγές αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βιετνάμ είναι περίπου ενός κύκλου εργασιών 40 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ήδη από τώρα το Βιετνάμ είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος και κάθε μέρα οι πολίτες μας χρησιμοποιούν προϊόντα made in Vietnam. Αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να βελτιώσει τις εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με ένα στρατηγικό εταίρο σε μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή όπως είναι η ε, Νοτιοανατολική Ασία σε ένα σύστημα ε, με σαφείς και κοινού κανόνες. Το Βιετνάμ τα τελευταία χρόνια έκανε μια πορεία πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων κυρίως όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα ε, και κυρώθηκαν και από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας τα όσα έγιναν σε εργατικό δίκαιο. Και φυσικά θα πρέπει να επιμείνουμε και σε αυτό και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ελευθερία έκφραση και να ζητήσουμε συγκεκριμένε πράξει ε, από πλευρά ε, Βιετναμέζικων αρχών. Γι' αυτό και η συμφωνία αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό μοχλό στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να πιέσει το Βιετνάμ να σεβαστεί τι δεσμεύσει που έχει αναλάβει. Ευχαριστώ, συνάδελφο Σαράντσοβα. Έχει τώρα το λόγο για ένα mm. λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αυτή θα είναι η πρώτη σημαντική εμπορική συμφωνία που το νέο κοινοβούλιο θα ακυρώσει και θα στείλει αρκετά θετικά μηνύματα με αυτό. Καταρχάς, σε αυξανόμενο προστατευτικό κόσμο πιστεύει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ελεύθερο εμπόριο βάσει κανόνων. Δεύτερον, στέλνουμε μήνυμα προς την περιφέρεια και πλησιάζουμε κατά ένα βήμα στην μια περιφερειακή συμφωνία με τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Μήνυμα προ του πολίτε και τι επιχειρήσει είναι το τρίτον, που θέλουμε να επιβάλλουμε καλύτερε συνθήκε για τι επιχειρήσει μα να μπορούν να ανθούν, να μεγαλώνουν και να δημιουργούν θέσει εργασία. Τέλο, αποδεικνύεται ότι το εμπόριο ε, επηρεάζει θετικά άλλου τομεί. Οι διαπραγματεύσει προώθησαν το Βιετνάμ προ σημαντικέ εργασιακέ μεταρρυθμίσει. Έχοντα αυτό το πλαίσιο, υπάρχει ένα τρόπο οικοδομικά να συνομιλήσουμε για θέματα που ποικίλουν από ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι περιβάλλον. Όπως με κάθε συμφωνία, η εφαρμογή θα είναι το κλειδί και μπορείτε να βασιστείτε στο Κοινοβούλιο ότι θα κάνει τη δουλειά του πάνω σε αυτό. Και ευχαριστώ. Καπομενόζη, για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χρησιμοποιούμε τα σωστά λόγια για να σχολιάσουμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψεύδι δεν θα δημιουργηθεί τοπική ανάπτυξη των βιετναμικών επιχειρήσεων, θα χρησιμεύσει μόνο να δώσει κίνητρα για μεταγκαταστάσεις των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και μεγάλων πολυεθνικών προς ε, μια χώρα όπως είναι το Βιετνάμ. Άλλο ένα πλήγμα λοιπόν για αυτό το τομέα που αποδημιουργήσει προβλήματα στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Ντροπή επίσης. Διότι το είπαν πολλοί, τα ανθρώπινα δικαιώματα σίγουρα δεν γίνονται σεβαστά στο Βιετνάμ, τα κοινωνικά πρότυπα είναι ελάχιστα και πολλαπλή εμπορική συμφωνία που θα ευνοήσει μια προς τα κάτω ε, κάτω ανταγωνισμό όσον αφορά το μισθολόγιο, υποκρισία, διότι το νέο πράσινο σύμφωνο που θέλετε να επιβάλλει τι επιχειρήσει μα και θα κοστίσει πάρα πολύ σε αυτέ, προφανώ δεν μπορεί να επιβληθεί στο Βιετνάμ και το Βιετνάμ θέλει να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση με πρότυπα που θέλετε υποτίθεται να ζητήσετε να εφαρμόζει η Μεγάλη Βρετανία που τα σέβεται τώρα. Λοιπόν, χρεοκοπημένη είναι η εμπορική σας πολιτική και συνάπτεται ε, συμφωνίες με απόμακρες χώρες που έχουν ε, πολύ τη χάρπα στα πρότυπα για τα εργαστικά δικαιώματα. Χάουταλα, έχετε λόγο για ένα λεπτό, Πρόεδρε, Επίτροπε. Οι συμφωνίε μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του Βιετνάμ αδιαμφισβήτητα είναι σημαντικέ συμφωνίε γεωπολιτικώ και το Βιετνάμ έκανε πρόοδο στι μεταρρυθμίσει για το εργασιακό δίκαιο, αλλά από την άλλη πλευρά πέτυχε να αλλάξει τον ποινικό του κώδικα, να επιτρέψει στου εργάτε να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα. Η καταστολή έγινε πιο σοβαρή ακόμα και στην τελευταία φάση ε, των συμφωνιών το Κοινοβούλιο, εάν δώσει τη σύμφωνη γνώμη του αύριο, ε, θα φέρει μεγάλη ευθύνη, διότι οι δικέ του απαιτήσει δεν μπορούν να υλοποιηθούν όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ανθρώπινα δικαιώματα και τη συμμετοχή μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών. Και όπω η Επιτροπή μα των Εξωτερικών Υποθέσεων απαιτεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ομολογή του στο Βιετνάμ, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό ανεξάρτητο εποπτεία όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και μηχανισμό υποβολή καταγγελιών και δυνατότητα ε, διορθωτικών ε, μέτρων και προσφυγών. Γι' αυτό η ομάδα μα οι πράσινοι, δεν μπορούν ακόμα να υποστηρίξουν αυτές τις συμφωνίες. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, Μπιέλαν. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και η Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών και η Επενδυτική Συμφωνία είναι πολύ φιλόδοξε, οι πλέον φιλόδοξε που έχει συνάψει με αναπτυσσόμενη χώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η διαπραγμάτευση ε, από πλευρά Κομισιόν επί δύο και δύο στόχου. Πρώτον, οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να έχουν ε, την καλύτερη πρόσβαση ε, στι αγορέ. Και το δεύτερο, ε, να είναι μετά τη Σιγκαπούρη, ένα δεύτερο σημείο αναφορά, το Βιετνάμ στην περιοχή αυτή. Και εκπληρώθηκαν, επετέχθησαν πλήρω αυτοί οι δύο στόχοι. Μάλιστα, οι δύο συμφωνίε ε, υπερβαίνουν και τι υποχρεώσει στο πλαίσιο του ΠΟΕΣ, το τομεί όπω υπηρεσίε, δημόσιε προμήθειε, μη δασμολογική φραγμή, ε, δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, γεωγραφικέ συνδείξει. Και σε όλου αυτού του τομεί ε, συμφωνεί το Βιετνάμ να αναλάβει νέε δεσμεύσει που υπερβαίνουν τα όσα προέβλεπαν άλλες συμφωνίες και ο, ε, η CPTPT. Με τις συμφωνίες αυτές όλοι οι θεσμολογικοί φραγμοί σχεδόν καταργούνται, είναι ισορροπημένε οι διατάξει και θα είναι θετικέ επιπτώσει για τι οικονομίε των δύο πλευρών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει περισσότερε δυνατότητε να ασκεί πιέσει στο Βιετνάμ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητώ λοιπόν να στηριχθούν αυτέ οι δύο συμφωνίε. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Τζέρι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι σήμερα συναντώνται τα άκρα. Αυτοί που είστε αντίθετοι σε αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να το σκεφτείτε διπλά. Ποιο είναι ο στόχο, Ο στόχο είναι να δημιουργηθούν κίνητρα και οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να επενδύσουν περισσότερο. Αυτέ οι εμπορικέ συναλλαγέ θα ευνοήσουν την ανάπτυξη ε, και τα πρότυπα και η δημοκρατία ε, θα επεκταθούν σε αυτή τη χώρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δίνουμε μαθήματα ε, στις άλλε χώρε. Ε, ουσιαστικά θέλουμε να δείχνουμε σεβασμό και να αναπτύσσουμε σχέσεις με τους γείτονε. Ο διάλογος, ε, η παρακολούθηση των εξέλιξεων θα βελτιώσουν την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τα εργασιακά κοινωνικά πρότυπα στο Βιετνάμ. Όσοι είναι κατά τη συμφωνία, δεν θέλουν να έχουν πρόσβαση ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, ε, στις ε, δημόσιες προμήθειες στο Χανό και στο Χονσιμί. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ο Επίτροπος θα μπορούσε να δώσει πρακτικές πληροφορίες, ώστε οι ΜΜΕ να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρω αυτό το δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Ροντρίγκεφ Πινιέρο τώρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Χόγκαν, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Βιετνάμ έχει πολύ μεγάλη στρατηγική σημασία λόγω τη όθηση που δίνει στι εμπορικέ μα σχέσει με την περιοχή τη ΑΣΕΑΝ και με την ε, σαφή δέσμευση του Βιετνάμ για να προστατεύσει ε, την βιώσιμη ανάπτυξη και την πολυμερή ανάπτυξη όταν το χρειαζόμαστε περισσότερο μειώνονται με φιλόδοξο τρόπο οι δασμοί και κυρίως υπάρχει ένα δεσμευτικό κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης που καθορίζει ένα πλαίσιο εργασιακών σχέσεων ε, που συνάδει περισσότερο με τις αρχές ε, του ε, ILO. Ε, χάρη στην όθηση της ε, κοινοβουλευτικής μου ομάδας αλλά και άλλων ομάδων καταφέραμε να έχουμε ε, παραχωρήσεις από πλευράς κυβέρνησης του Βιετνάμ σε θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων κυρίως σε θέματα εργασίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που έγιναν ε, από πλευρά ε, αρχών του Βιετνάμ. Αλλά απομένουν ακόμα πολλά και εμεί οι σοσιαλιστέ και δημοκράτε ανησυχούμε ιδιαίτερα όσον αφορά τα ε, θεμελιώδει ελευθερίε. Θα παρακολουθούμε στενά λοιπόν την εφαρμογή τη συμφωνία και θα ήθελα να ζητήσω, κύριε Επίτροπε, να λάβετε και τα απαραίτητα μέτρα για να μα εξασφαλίσετε ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι ει βάρο των Ευρωπαίων Γεωργών και κυρίω των παραγωγών ρυζιού. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για να προχωρήσουμε η συμφωνία και θα την υποστηρίξω. Ευχαριστώ. Κάρλε Κίντ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συναδελφοί, θα ήθελα να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Μπαρτόλο που ήταν εισηγητής για την Επιτροπή Αλίας ε, για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Η καταπολέμηση της παράνομης αλίας σημαίνει ότι θα έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη των πόρων και επίσης θα αποφύγουμε και τον αθέμητο ανταγωνισμό από αλίες που δεν ε, ε, τηρούν τις δεσμεύσεις που έχουμε και εμείς στην υπηρή μας. το Βιετνάμ λοιπόν έχει κάτι για την παράνομη αλία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι προσπάθειε που έκανε η χώρα αυτή, στα πλαίσια τουλάχιστον των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν σήμερα σε αυτή τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Επίση, στη συμφωνία αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα συμβαλόμενα μέρη θα δώσουν ενεργό μάχη κατά τη παράνομη αλεία. Ε, αρκεί αυτό. Ε, αν δεν είναι αρκεί, τότε να πάμε πιο πέρα και να ζητήσουμε, για παράδειγμα, και άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα ε, την κατάργηση των προτιμησιακών δασμών για την αλληλεία και ότι στο μέλλον θα δώσουμε κίτρινη κάρτα. Αυτή την τροπολογία υπέβαλε το ΡΙΝΙΟΥ γι' αυτό το λόγο και θα ήθελα να σας ζητήσω να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ, Σνάφος Κράχ, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το εμπόριο ε, θα βοηθήσει και τις δύο πλευρές σημαντικά. Είμαι ε, μόνιμος ηγητής για τον Μπαγκλαντές και άλλα κράτη και γνωρίζω πολύ καλά ε, ότι οι αναψώμενες χώρες βλέπουν το Βιετνάμ θετικά. Βλέπουν τι μπορεί να αποκομίσει από μια εμποριακή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι μπορεί αυτό να το βοηθήσει να αναπτυχθεί. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι σημαντική αυτή η συμφωνία για τις πολλές αναπτυσσόμενες χώρες προσφέρει, αναδυόμενες χώρες προσφέρει δυνατότητες και γι' αυτό θα ζητήσω την υποστήριξη αυτή της ισορροπημένης συμφωνίας που λαμβάνει υπόψη τις διάφορες ε, απόψεις ε, ε, στο σώμα για τις εμπορικές σχέσεις με τρίτες χώρες και νομίζω ότι είναι μια προσφορά ανάπτυξη σε μια αναδυόμενη χώρα ώστε και τα άτομα αυτά να παραμένουν στη χώρα τους και να μην αναζητούν την τύχη τους σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι είναι λοιπόν μια ισορροπημένη συμφωνία που ρίχνει ένα θετικό φως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα την υποστηρίξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος Γκρεγκόροβ έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ. Το ελεύθερο εμπόριο εν γέννη δημιουργεί πλούτο και για τις δύο πλευρές. Σαν Ευρωπαία. πώς μπορώ να είμαι κατά μιας τέτοιας συμφωνίας επειδή δίνουμε λευκό κάρτα σε ένα αυταρχικό καθεστώς για να ε, έχει εμπορικές σχέσεις με τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο χωρίς να έχουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Κυρώντας αυτή τη συνθήκη λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξει μια χώρα όπου έχει ένα και μοναδικό κόμμα, μετά από ένα μοναδικό κόμμα που καταπιέζει τον κόσμο. μη γελιέστε από τι εγγύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι ε, δημοκρατικέ μεταρρυθμίσει που υπόσχονται. Τα 8 χρόνια των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία αυτή, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στο Βιετνάμ. Δεν είναι μόνο το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, θα ήταν κάτι που θα ήταν ε, δυσμενέ και για το εμπόριο. Έχει πολλά περισσότερα να κερδίσει το Βιετνάμ από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη συμφωνία. Και τέτοιε στιγμέ θα πρέπει να έχουμε εγγυήσει όσον αφορά την πολιτική που ακολουθείται και τι επιχειρήσει μα. Θέλουμε μια Ευρώπη η οποία να μπορεί να επηρεάζεται από τα αυταρχικά καθεστώτα χωρί να δείχνουν σημάδια βελτίωση. Ευχαριστώ. Δέχεστε μια μπλε κάρτα από τον συνάδελφο Σίμων. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν κατάλαβα πολύ καλά τα επιχειρηματά σας. Πιστεύει ότι με ή χωρίς τη συμφωνία μπορούμε να έχουμε περισσότερη επιρροή σε αυτό το αυταρχικό καθεστώς. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα.